Please sit down. I think we can start. First of all, it is a one... Σκαθίστε συναδελφοί να ξεκινήσουμε. Ε, χαίρομαι πολύ που καθόμαστε εδώ δίπλα-δίπλα με τον Brian Simpson. Ήταν Πριν ε, καιρό που τον είδαμε τελευταία φορά, ελπίζω ότι είναι καλά. Ε, ε καλώς ορίσατε κύριε Σίμψον στην Επιτροπή Μεταφορών. Και τώρα μετά από αυτά τα ωραία αγγλικά ξεκινώ στα γερμανικά. Ε, τα αποτελέσματα από του συνεδρίε των συντονιστών σήμερα το πρωί έχουν μοιραστεί τα αντίτυπα. Αν δεν υπάρχουν προβλήματα μέχρι τις 5.30 το απόγευμα σήμερα θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται. Μετά, Πάμε στην ψηφοφορία για τη συμφωνία για την ε, τροποποίηση του κανονισμού για την συλλογή δεδομένων ε, για τα ατυχήματα. Εισηγητή ο κύριο Κράμερ, φαντάζομαι ξέρετε ποιο είναι. Ψηφίζουμε λοιπόν. Να ελέγξουμε πρώτα ηλεκτρονικά το σύστημα. Άρχεται η ψηφοφορία. Όλα εντάξει. Δεν έχουμε υπεράριθμους. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Abstimmung ist Πέρας ψηφοφορίας. 34 ψηφίσατε, 32 υπέρ, 2 αποχές, καμία ψήφος κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην ψηφοφορία... Α, όχι. Πάμε στην ανταλλαγή απόψεων με τον Brian Simpson, τον Ευρωπαίο συντονιστή για, τους, ε, για τις θαλάσσιες ε, διόδους. Ε, θα μας κάνει μια ανακοίνωση για τους Motorways of the Sea. Όχι για τους σιδηροδρόμους αυτή τη φορά. Έχεις 10-15 λεπτά. Brian, σε ακούμε. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συγγνώμη, συνάδελφοι, αλλά εφόσον είναι εδώ ο Μπράιαν, καταλαβαίνετε, πρέπει να κάνετε λίγο ησυχία. <laughs> Well, thank you very much, uh, Ευχαριστώ, Μάικλ, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι για τα πολύ καλά σας λόγια, για την θερμή σας υποδοχή. Κυρίες και κύριοι, είμαι σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσω το λεπτομερές εφαρμοστικό σχέδιο για τους διάβλους της θάλασσας. Είναι το πρώτο μου πρόγραμμα εργασίας που καταγράφει το όραμα για το μέλλον των διάβλων της θάλασσας ως τμήμα της, της θαλάσσιας διάστασης του TEN-T, του Διευρωπαϊκού Δικτύου. Η Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά το δικτύο TEN-T, οπότε δεν θα επικεντρωθώ σε γενικά σχόλια για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ε, μεταφορές, ε, ούτε τις προκλήσεις και τους στόχους της. Θα ήθελα απλώς να χρησιμοποιήσω τα επόμενα 10-15 λεπτά για να σας καθοδηγήσω σε αυτό το συνολικό έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει την, ε, το λεπτομερές εφαρμοστικό σχέδιο. Για να ξεκινήσω, θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντική είναι η πολιτική αυτή για τη συνολική ενσωμάτωση, ολοκλήρωση των ε, ε, διαδρόμων μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή, αυτός ο όρος ε, αναφέρεται νομικά και περιγράφεται στο άρθρο 21 του κανονισμού TEN-T 1315 του 2013 και ονομάζεται οι κατευθυντήρες γραμμές της Ένωσης για την εκπόνηση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Σύμφωνα με τούτο τον κανονισμό, οι διάβλοι της θάλασσας θα πρέπει να βοηθήσουν στην επίτευξη του ευρωπαϊκού χώρου θαλασσίων μεταφορών χωρίς εμπόδια. Είναι λοιπόν μια οριζόντια διάσταση της ευρωπαϊκής πολιτικής για, την, για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Ε, μια πολύ σημαντική διάσταση είναι η, διάσταση του τέντη στη συνολική πολιτική. Γιατί χάρη στην, ε, στις μεταφορέ, μεταφορές εξασφαλίζουμε 40% του εσωτερικού εμπορίου και 75% του εξωτερικού εμπορίου ε, μετακινώντα αγαθά και άτομα από τις θαλάσσιες οδούς μπορούμε να αποφύγουμε την συμφόρηση ε, στις, στις χερσαίες οδούς και να έχουμε και οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά ωφέλη. Προφανώς, η θαλάσσια πολιτική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην δημιουργία διασυνδέσεων μεταξύ της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τρίτων χωρών. Έχουμε στην Ευρώπη πάνω από 800, 800 ε, ε, συνδέσεις ε, ρορό και εμπορευματοκιβωτίων. Ε, χρησιμοποιούνται πάνω από 400 λιμένες και συνδέουν ε, εκατοντάδες ε, λιμένες παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι το 2014 οι ευρωπαϊκοί λιμένες διαχειρίστηκαν 3,8 δισεκατομμύρια τόνους κάργο. Περίπου 3 δις τόνοι είναι ε, όγκος που που μεταφέρθηκε από τις ε, ε, θαλάσσιες, από τις, συγγνώμη, από τις χερσαίες μεταφορές ή τις υδροδρομικές μεταφορές στην θαλάσσια. 79 ευρωπαϊκοί λιμένες βρίσκονται σε σύνδεση με έναν από τους εννέα βασικούς διάβλους, χερσαίους διάβλους. Και αυτό σημαίνει δύο τρίτα της συνολικής κίνησης στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Τώρα, για το θέμα της ανάπτυξης. Τα ευρωπαϊκά, οι ευρωπαϊκοί λιμένες συνδέονται άμεσα με πάνω από 800.000 επιχειρήσεις. Συνολικά καλύπτονται 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Μονατέθηκε ο ρόλος αυτός του Ευρωπαίου ε, συντονιστή για τις ε, θαλάσσιες διάβλους. Μπορεί κάποιοι να ήσασταν ε, παρόντε ε, όταν μου αποδόθηκε η ευθύνη αυτή πριν την λήξη τη προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Ο κανονισμό Τεντή ε, προβλέπει ότι εντό δύο, χρόνων ε, μετά, την δική μου, μετά το δικό μου διορισμό θα πρέπει να σα παρουσιάσω ένα λεπτομερέ εφαρμοστικό σχέδιο με βάση τις εμπειρίες που έχουμε που σχετίζονται με, τις, με τη θαλάσσια πολιτική της Ένωσης. Και γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ σήμερα για να σας ε, παρουσιάσω αυτό ακριβώς το σχέδιο. Το έγγραφο αυτό βεβαίως είναι η αρχή μόνο. Η δική σας συμβολή αλλά και η συμβολή των κρατών μελών και των εμπλεκόμενων φορέων είναι απαραίτητη για να εμπλουτίσουμε το κείμενο αυτό και να ορίσουμε τον, τις δράσεις και την ε, στοχοθέτηση των θαλασσίων λεωφόρων. Μόλις έχει γίνει και ολοκληρωθεί αυτή η διαβούλευση, θα υπάρξει πιο σαφής και λεπτομερής καθοδήγηση για το μέλλον της πολιτικής για τις θαλάσσιες λεωφόρους. Ε, με άλλα λόγια, θα πρέπει να δούμε προς τα, ποιου ε, προς τα θα πρέπει να ε, προσανατολιστούμε και ποια είναι τα μέσα που θα υπάρχουν στη διάθεσή μας. Περί τίνος πρόκειται λοιπόν. Το έγγραφο αυτό έχει τρεις βασικούς πυλώνες για την ε, ναυσιπλοεία και τα ε, λιμάνια, τα οποία, τους οποίους έχω θεωρήσει εγώ ως βασικές προτεραιότητες. Μία είναι το περιβάλλον. Μία είναι η ενσωμάτωση της ε, θαλάσσιας μεταφορά, των θαλασσιών μεταφορών στην αλυσίδα επιμελητίας και η θαλάσσια ασφάλεια, διαχείριση κίνησης και το ανθρώπινο στοιχείο, ο ανθρώπινος παράγοντας. Το 2016 έγινε μια ε, ευρεία διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κράτη-μέλη και με εσάς, τους ε, ευρωβουλευτές. Ε, οργάνωσα τρεις συναντήσεις, τρία φόρουμ, τον Μάρτιο και τον Μάιο, με τις, όπου συζητήθηκαν οι συγκεκριμένες προτεραιότητες. Για ποιο λόγο έγιναν όλες αυτές οι συναντήσεις. Θέλαμε να έχουμε όσο δυνατόν πιο, α, πιο απαντήσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς για το ποιοι είναι οι τομείς όπου θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις θαλάσσιες λεωφόρους. Και βεβαίω θα πρέπει να δούμε και τον σχετικό προπολογισμό. Το έγγραφο που σα παρουσιάζω σήμερα αποτελεί μια περίληψη όλων αυτών. Και να τονίσω, παρακαλώ, ε, δώστε μου την ευκαιρία, τα πιο βασικά σημεία του. Για την πρώτη προτεραιότητα, το περιβάλλον. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό τομέα και αξίζει τον κόπο να σημειώσουμε ότι η ε, βιομηχανία θαλασσίων μεταφορών είναι η μόνη που έχει, έναν, που έχει κανονισμό για τις ε, εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα οι θαλάσσιες λεωφόροι μπορούν να βοηθήσουν για να υπάρξει καλύτερη συμμόρφωση με την ε, νομοθεσία και θα πρέπει να προωθήσουν project που να σχετίζονται με την ε, ποιότητα του αέρα, να βοηθήσουν τη βιομηχανία να συνάδει με τις ε, εκπομπές για την ποιότητα του αέρα και με τη ΣΕΚΑ, τον, τις, για το σημείο ελέγχου δηλαδή της, των εκπομπών θείου. Επίσης, να υπάρξει καλύτερη ανάπτυξη του υγροποιημένου φυσικού αερίου και της χρήσης της μεθανόλης ως και άλλων τεχνολογικών ε, επιλογών. Και επίσης να δούμε πώς μπορούμε να, ε, να διαχειριστούμε την αποθήκευση υγροποιημένου αερίου και να βελτιώσουμε την ε, αποτελεσματικότητα και τη μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων για να μειώσουμε τις, το αποτύπωμά μας σε εκπομπές οξυδιού του άνθρακα. Επίσης, για την επιχειρησιακή μόλυνση θέλουμε να έχουμε καλύτερα συστήματα για τη διαχείριση νερών στα σκάφη, ανακύκλωση κτλ. Okay, Επίσης πρέπει να δούμε την ε, μόλυνση μετά από ατυχήματα. Πρέπει να δούμε καλύτερα μέτρα ασφαλείας και κατάρτισης ε, που είναι απαραίτητα για να βελτιώσουμε τα παγκόσμια επίπεδα ασφάλειας και να ε, απαλύνουμε την, ε, τις, ε, επιπτώσεις των, της μόλυνσης που προέρχεται από ατυχήματα. Και επίσης η πράσινη ναυσιπλοεία και τα μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Δεύτερος πυλώνας είναι η ενσωμάτωση της, των φαλαισίων μεταφορών στην λυσίδα επιμελητίας. Ο δεύτερος αυτός πυλώνας έχει να κάνει με την με, αυτή ακριβώς, με αυτό ακριβώς το θέμα και οι θαλάσσιες λεωφόροι αποτελούν πολύ σημαντικό τομέα για να συμβάλλουν στην αποτελεσματική πολιτική έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές. Ε, πρέπει λοιπόν να έχουμε αποτελεσματικούς, αποτελεσματικές διάβλους που θα συνδέουν και τα, τα πλοία με τους ε, χερσαίους διάβλους. Οι λύσεις βεβαίως είναι πολλές και μπορούν να εφαρμοστούν και για τις θαλάσσιες και για τις χερσαίες μεταφορές. Υπάρχουν πολλές ε, φιλοδοξίες και πολλές ε, ε, απαιτήσει για να βελτιωθούν τα πράγματα. Πρέπει να ε, έχουμε καλύτερες ε, υπηρεσίες διαχείρισης ε, για να μπορέσουμε και στην ξηράδα και στα σκάφη να διαχειριστούμε καλύτερα τις ροές κίνησης. Επίσης, πρέπει να βελτιώσουμε τις συνδέσεις προ τα λιμάνια και να ε, προωθήσουμε την, τον συγχρονισμό και την διαφοροποίηση των πηγών μεταφορών. Πρέπει να υποστηρίξουμε την ανταλλαγή πληροφοριών έτσι ώστε τα ε, σκάφη να μπορούν να ανταλλάσσουν μέσω των καλύτερων δυνατών συστημάτων πληροφορίες για να μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τις ε, υπηρεσίες τους αλλά και να είναι πιο αποτελεσματικές οι διαδικασίες cargo στις ε, υπερπόντιες περιοχές που ξέρω ότι πολλοί ε, από εσά τους ενδιαφέρουν. Οι θαλάσσιες λεωφόροι μπορούν να υποστηρίξουν τη σύνδεσή τους με την ε, ενδοχώρα για να μην ξεχαστούν στην όλη πολιτική τέντη και να ενισχύσουν το γεωστρατηγικό δυναμικό των νησιών προωθώντας ας πούμε της, τη δυνατότητα ύπαρξης σταθμών για την χρήση του υγροποιημένου αερίου. Επίση, η θαλάσσια ασφάλεια, η διαχείριση είναι ο τρίτος πυλώνας του σχεδίου μας. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ διαφόρων στοιχείων, ασφάλεια στη θάλασσα, ασφάλεια στο λιμένα, διαχείριση της κίνησης και κατάρτιση, που βεβαίως έχει να κάνει με το ανθρώπινο στοιχείο. Το ε, λεπτομερές ε, εφαρμοστικό σχέδιο αποτελεί, ε, περιλαμβάνει συγγνώμη, έναν ε, μεγάλο αριθμό στόχων που βεβαίως θα πρέπει να ε, επιτευθούν στα πλαίσια του προγράμματος των θαλασσίων λεωφόρων. Για την ασφάλεια πρέπει να έχουμε σωστό προγραμματισμό και να κάνουμε διάφορες δοκιμές για να αντιμετωπιστούν ε, ε, περιπτώσεις εκένωσης ή ε, επίγουσας κατάστασης. Για τα κρουαζιερόπλια για παράδειγμα. Το ανθρώπινο στοιχείο, να μειώσουμε τον κίνδυνο που υπάρχει από το ανθρώπινο λάθος, να προωθήσουμε διατομεακές, διατομεακά προσόντα και να μπορέσουμε να έχουν, ή, ε, να έχουν τα πληρώματα μια συνολική άποψη για να ξέρουν ποια είναι ακριβώς, ή, ποιες είναι ακριβώς οι διαδικασίες ασφάλειας πάνω στο πλοίο. Και επίσης πρέπει να έχουμε νέα προσέγγιση για την κατάρτιση για τις νέες τεχνολογίες, για παράδειγμα για το υγροποιημένο αέριο. Ε, διαχείριση ε, κίνησης. Πρέπει να υπάρξει ένα maritime ICT, να υπάρξει ψηφιοποίηση και συστήματα θαλασσίων, ε, ανταλλαγής πληροφοριών θαλασσίων μεταφορών. Επίσης να υπάρχουν πλατφόρμες ανταλλαγής τέτοιων πληροφοριών, να υπάρχει καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην, στις παραδοσιακές, στο παραδοσιακό σύστημα πληροφορικής με βάση τους καπετάνιους και με βάση τους, τα συστήματα που υπάρχουν στην ενδοχώρα. Επίσης, πρέπει να αναλάβουμε δράσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από τον προπολογισμό για τις θαλάσσιες λοφόρους. Το έγγραφο που σας έχω υποβάλει είναι πλήρες και περιλαμβάνει μια σειρά πιθανών δράσεων που βασίζονται σε αυτούς ακριβώς τους τρεις πυλώνες που σας ανέφερα περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων και καλύπτει ένα πλήρες φάσμα πιθανών ε, επιλογών σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του τέντη. Οι επόμενοι 12 μήνες ε, των διαβουλεύσεων θα πρέπει να μας ε, δώσουν τη δυνατότητα να περιορίσουμε τον αριθμό αυτών των δράσεων, οπότε, οπότε οι θαλάσσιες λεωφόροι θα, θα μπορέσουμε να τις οργανώσουμε καλύτερα και στο μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο. Εγώ θα εμπλακώ στενά με, σε διάλογο με τα κρατημέλη, με το Ευρωκοινοβούλιο και με τους εμπλακόμενους φορείς για να μπορέσουμε να χτενίσουμε καλύτερα τις πιο σημαντικές ε, δράσεις ε, που θα χρηματοδοτηθούν από τον ε, προπολογισμό μας. Κάποια από τα κεφάλαια αυτού του κειμένου έχουν να κάνουν με την συλλογή δεδομένων. Θέλω να συλλέξουμε όλα τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα για τα, και για τους λιμένες στην Ευρώπη, να δούμε ποιες είναι, ποιοι είναι οι βασικοί δείκτε απόδοση και να δούμε πού υπάρχουν κενά. Αν μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, συμμόρφωση με την παραβολητική, με την ε, πολιτική και έτσι θα, να μπορέσουμε να είμαστε στη θέση να προτείνουμε πιο στοχοθετημένες δράσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από τον μελλοντικό προπολογισμό για τις θαλάσσιες λοφόρους. Τώρα, δύο, ε, δύο λόγια για τη χρηματοδότηση. Μέχρι τώρα το TEN-T και το SEF έχουν επενδύσει στην πολιτική θαλασσίων λεωφόρων 651 εκατομμύρια ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Το δεύτερο ΣΕΦ του 2015 εξεκολουθεί να τρέχει. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε δύο μέρες. Αλλά ο συνολικός του προϋπολογισμός έφτανε τα 280 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 150 εκατομμύρια ευρώ θα αποδοθούν στις χώρες συνοχής. Είναι σημαντική λοιπόν η στήριξη αυτή, αλλά έχοντας υπόψη ότι οι θαλάσσιες λεωφόροι είναι οριζόντια προτεραιότητα και περιλαμβάνει τόσο πολύ μεγάλο δυναμικό, δεν είναι αρκετός ο προπολογισμός αυτός. Μέχρι τώρα η εφαρμογή του ΣΕΦ δείχνει ότι υπάρχει υπερ Υπάρχει υποαπορρόφηση του προπολογισμού και μάλιστα πολλοί από τα προγράμματα που θα άπτοντον, που θα άπτοντο των ε, θαλασσίων ε, λεωφόρων ε, χρειάστηκε να απορριφθούν. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε ένα, μια αναθεώρηση του πολιετούς χρηματοοικονομικού πλαισίου και να εξασφαλίσουμε ότι η σημασία των, της πολιτικής των θαλασσίων λεωφόρων θα αντικατοπτρίζεται σωστά και σε ό,τι αφορά τις πολιτικές προτεραιότητες και, στον, και στα κονδύλια που θα α, αποδοθούν σε αυτή. Τα κονδύλια του ΣΕΦ αποτελούν βεβαίω ένα σημαντικό στοιχείο για να ε, συνδεθούν οι θαλάσσιες λεωφόροι με το τέντι και το σχέδιο εφαρμογής θα αποτελέσει ένα ε, καλό ε, έναυσμα για να, υπάρξει, να υπάρξουν αξιόλογα project στα πλαίσια του, των θαλασσίων λεωφόρων αλλά και στι στις μελλοντικές, στους που θα γίνουν για το ΣΕΦ. Ζητώ λοιπόν από τα μέλη της Επιτροπή σα τη στήριξη και για το πρόγραμμα μου αλλά και για τις θαλάσσιες λεωφόρου συνολικά όταν θα έρθει η στιγμή να ξεκινήσετε να συζητάτε τις, ε, τους, τον Το έγγραφο αυτό είναι μείζων σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη της, ε, των θαλασσίων μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά δεδομένα που σχετίζονται με τις θαλάσσιες ε, λεωφόρους έχουν συλλεγεί μέχρι τώρα, είτε μέσω ε, εμπειρία που έχουμε, είτε μέσω project που είτε ολοκληρώθηκαν είτε τρέχουν ακόμη. 80 τον αριθμό. Επίσης, συλλέγουμε πολλές πληροφορίες και από ε, συζητήσεις που κάνουμε με τους ε, εμπλεκόμενους φορείς, ε, με τον κλάδο, με τα κρατημέλη. Το λεπτομερές εφαρμοστικό σχέδιο αντικατοπτρίζει διάφορες απόψεις και αποτελεί τη βάση για ένα συνεκτικό πρόγραμμα εργασίας που θα δίνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μαζί με τα υπόλοιπα άλλα προγράμματα εργασίας για τους εννέα στρατηγικούς πυλώνες για τα δίκτυα για τις λεωφόρους. Ε, τέλος, δίνουμε πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία στο TNT, συνολικά στα πλαίσια της ε, θαλάσσιας πολιτικής. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. να σας ε, δώσω το σχέδιο το σχέδιο εφαρμογής. Θα σας υποβάλω το σχέδιο αυτό εφαρμογής και είμαι σίγουρος ότι θα το έχετε διαβάσει μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Μεγάλη μας χαρά που σας ακούσαμε. Γιατί έχετε μεγάλη πείρα, 25 ετή πείρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό φαίνεται. Σας ευχαριστώ. Τώρα για τους ομιλητές, ο κ. Βαντερκάμπ. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό να βρούμε τα ακουστικά μας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν ένα διαδικαστικό ζήτημα που θα ήθελα να θίξω. Φαίνεται ότι η έκθεση του κυρίου Σίμψον έχει ε, διανεμηθεί ηλεκτρονικά. Δεν έχουμε όμως ε, αντίτυπα αυτού του βιβλίου. Έχουμε ένα άλλο έγγραφο, το δείχνει ο μιλητής, αλλά όχι την έκθεση του κυρίου Σίμψον. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να μου αποστείλετε ένα αντίγραφο, γιατί τουλάχιστον εγώ δεν το έχω λάβει. Θα προτιμούσα να έχω ένα αντίτυπο επιχάρτου ή δυνατόν. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον κύριο Σίμψον για την εργασία του. Η βιωσιμότητα είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, πολύ σημαντικό θέμα και θα ήθελα να μου πείτε γενικότερα πώς εντάσσεται η εργασία σας στον IMO. Ακούσαμε πολλά σε σχέση με την βιωσιμότητα και τον Διεθνή Οργανισμό Θαλασσίων Μεταφορών. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Τώρα το δεύτερο αφορά τις θαλάσσιες αρτηρίες και πώς εντάσσονται με άλλους τρόπους μεταφοράς, δηλαδή πώς ορίζεται η διατροπική μεταφορά, γιατί μιλήσατε και για μεταφορές ε, στην ενδοχώρα. Πώς συνδέονται οι δύο τομείς γιατί ε, πολλές φορές μιλάμε για το λιμάνι της Κωνσταντσα και για άλλες ε, ποτάμιες οδούς. Άμα μεταφερθεί κανείς, θέλει δηλαδή να περάσει από τη Βιέννη στην Κωνσταντσα, θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια μεταφοράς και αυτό αφορά και τα πληρώματα πάνω στο πλοίο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε κάτι να μας πείτε για την έλλειψη πληρωμάτων, γιατί πολλοί ε, ασχολούνται, απασχολούνται σε αυτό το τομέα σχετίζεται με τις πολυτροπικές μεταφορές τις οποίες ε, αναφερόμαστε. Είναι μια πολύ καλή απασχόληση. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ε, θέμα επαρκών πληρωμάτων. Επίσης, δεν γίνεται λόγος για επενδύσεις στις υποδομές, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πότε θα λάβουμε χρήματα για να προβούμε σε εργασίες υποδομών στους λιμένες. Και πώς αυτό συνδέεται με το CEF, συνδέοντας την Ευρώπη και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Δεν ξέρω κατά πόσο η χρηματοδότηση του ΕΦΣΥ θα επιλεγεί για τις ε, επενδύσεις αυτές. Αυτά ως προς το ΣΕΦ και το ΕΦΣΥ. Μιλήσαμε και στους συντονιστές για αυτό το θέμα, άρα νομίζω ότι αφορούν όλους και όχι μόνο εμένα. Ισμαήλ Ερτούκ, ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε, Μπράιαν, ξανά εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Και βεβαίω σε βάλαμε να καθίσει εκεί που έχει συνηθίσει κιόλα, έτσι. Σε ευχαριστώ για την ε, έκθεσή σου. Όσοι ήταν παρόντε εδώ στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο θα θυμούνται πόσο δύσκολο ήταν να μπουν σε λειτουργία αυτές οι motorways of the sea, αυτές οι θαλάσσιες αρτηρίες. Είχαμε δώσει εμείς υποστήριξη τότε, θυμούμε είχαμε και την εισηγήτρια εμείς, αλλά δεν ήταν σίγουρο εάν τελικώ θα υλοποιηθούν. Τώρα βλέπουμε όμως ότι η ιδέα ήταν καλή και όχι μόνο καλή. Ήταν και πραγματικά μια απόφαση στραμμένη στο μέλλον. Έχω δύο ερωτήσει. Αν θυμούμε καλά, είχαμε βάλει κάποιους φιλοδοξότερους στόχους τότε για αυτούς τους αυτοκινητόδρομους της θάλασσας, το πω έτσι, τις θαλάσσιες αρτήριες. Πότε θα μπορέσεις να μας δώσεις συγκεκριμένα νούμερα. Δηλαδή, εξοπλισμός για παράδειγμα με λιμάνια LNG, δηλαδή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Πότε θα έχουμε κάποιες απαντήσεις από τις χώρες μέλη και μια σύνοψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το που βρισκόμαστε. Δεύτερο, αν εξετάσουμε τις διάφορες αυτές διαδρομές, βλέπουμε ιδίως στις νότιες, Orient East, αλλά και τις βόρειες, στην Βαλτική. Είναι δηλαδή αυτές θαλάσσιες αρτηρίες που δραστηριοποιούνται σε γεωγραφικές περιοχές όπου έχουμε και αυτά τα σημαντικά προσφυγικά ρεύματα. Μέχρι τώρα έχει υπάρξει κάποια σύγκρουση με τους στόχους των θαλάσσιων αρτηριών. Δηλαδή, οι δύο αυτέ κινήσεις έχουν έρθει σε κάποια σύγκρουση και πώς σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος Κράμερ. Πριν να συνεχίσω τώρα, σας δείχνω αυτό το φυλάδιο, το οποίο επειδή είναι χοντρό και βαρύ δεν μπορούσε να διανεμηθεί. Σας έχουμε στείλει το link. Θα προσπαθήσουμε βέβαια και να το τυπώσουμε για να σα το στείλουμε. Αλλά το link σα το έχουμε δώσει. Και μην ξεχνάτε ότι είμαστε paperless. Είμαστε χωρίς χαρτί. Εγώ σας είπα πάντοτε ότι δεν είμαι paperless. Καμιά φορά βρίσκεσαι στη μειοψηφία. Ρόμπερτ Ευχαριστώ. Και εγώ χαίρομαι που ξαναβλέπω τον Μπράιαν. Καλώ ήρθε, Όπως πάντοτε ήσουν καλοδεχόμενο εδώ. Ευχαριστώ για την ε, πολύ σημαντική αυτή η έκθεση βέβαια. Εγώ δεν έχω μπροστά μου αυτά που έχει ο Μιχαήλ Κράμερ. Αλλά θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Και η πρώτη είναι σχετική με την ευθυγράμμιση με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης. Εκεί στην σελίδα 53 λέει input per barrier. Αλλά είναι λέει ουδέτερη σε ό,τι αφορά τη σχέση με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα. Είπε και για την διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη ότι ορισμένα χρήματα θα, θα ληφθούν από το σχέδιο Junkers. Βλέπεις κάποια συνέργεια μεταξύ του σχεδίου στρατηγικών επενδύσεων Junckers και τη στρατηγικής για τις θαλάσσιε αρτηρίες. Δεύτερο, γεωγραφική ερώτηση. Πού υπάρχει η καλύτερη σώρευση δυνατοτήτων για τις θαλάσσιες αρτηρίες και τη χρηματοδότησή τους. Λειτουργεί κάπου σε κάποιες χώρες καλύτερα από κάπου αλλού. Και πού υπάρχει η υψηλότερη ζήτηση για τις διασυνδέσεις αυτές των θαλάσσιων αρτηριών. Ενώ ίσως αλλού υπάρχει λιγότερη ανάγκη, λιγότερη χρήση δηλαδή θαλάσσιων αρτηριών. Γκεζίνε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Μπράιαν, για την έκθεσή σου. Όλοι όσοι σε γνωρίζουμε από προηγούμενες θητείες, ξέρουμε τι συμπαθητικός τύπος είσαι και ξέρουμε ότι κάνεις κάτι δουλειά. Και οι άλλοι που δεν σε ξέρουν τόσο καλά, θα σε μάθουν. Είμαι βεβαία. Τώρα, για τις δύσκολες ερωτήσεις που έχω να σου κάνω. Πάντως, κοίταξε, νομίζω ότι καλό ήταν που μας έδωσες τις προτεραιότητες για τη δουλειά σου. Έχω και κάποιες ερωτήσεις ακόμη. Δηλαδή, εγώ διαρωτώ με πάντοτε ποιο μπορεί να είναι ο ρόλο ενό συντονιστή σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Εσύ είπε, θα προσπαθήσει να προωθήσει, για παράδειγμα, την βιωσιμότητα. Έχω τώρα τρία θέματα. Το ένα είναι ότι και στην Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική και στην ε, Γύρω τη Μεγάλη Βρετανία έχουμε ποσοστά εκπομπών που πρέπει να γίνονται σεβαστά. Γι' αυτό και έχουμε ε, σκάφη που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Αυτή την περιορισμό δεν τον έχουν σε άλλες θάλασσες. Τα είχαμε συζητήσει την προηγούμενη περίοδο αυτά τα πράγματα, διότι σημαίνουν στρέβλωση του ανταγωνισμού. Τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό. Δεύτερο, πάλι υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG. Μπορείς με κάποιο τρόπο να ασκήσεις πίεση ώστε να χρησιμοποιηθεί περισσότερο. Έχουμε και αυτή την alternative fuel strategy μέχρι το 2020 υποτίθεται θα την υλοποιήσουμε. Αρχικά πήγαινε γρηγορότερα. Στο μεταξύ έχει πέσει τόσο πολύ τιμή του πετρελαίου που δεν υπάρχει πλέον κίνητρο. Εσύ τι μπορείς να κάνεις για να έχεις κάπως θετική ανταπόκριση. Τέλος πάλι για το περιβάλλον άκουσα πρόσφατα ότι υπάρχουν λιμάνια τα οποία δεν έχουν επαρκείς ε, δυνατότητες για δέσιμο σκαφών και για την ε, αποχέτευση των ε, βρώμικων νερών του σκάφους. Τι μπορείς να κάνεις εκεί. Τέλος. National Single Window και αλυσίδες εφοδιαστικής. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα έχουν όλα τα λιμάνια από το 2015. Δεν τα έχουν εφαρμόσει όμως όλες οι χώρες μέλη. Πάλι εκεί ως συντονιστής πόσο μπορείς να υψώσεις τη φωνή σου και να πιέσεις ώστε να αρχίσουν επιτέλους να τα εφαρμόζουν. Είχαμε κάνει σχετική έκθεση και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτε μέγα πρόβλημα. Βεβαίω και για την ε, ψηφιοποίηση και για τη διευκόλυνση των ε, εμπορικών οδών. Ακόμα δύο ερωτήσει. Πρώτον, εκπαίδευση. Μίλησε ότι είναι σημαντικό αυτό, η εκπαίδευση δηλαδή, για την ασφάλεια. Τι επιρροή μπορεί να ασκήσει ο συντονιστή στα σχολεία του εμπορικού ναυτικού δηλαδή. Μέχρι τώρα δεν έχω δει να εντάσσεται αυτό στι θαλάσσιε αρτηρίε. Βεβαίω χρειάζεται προσωπικό και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό στα ποντοπόρα πλοία. Τι, μπορείς, τι επιρροή μπορεί να ασκήσει λοιπόν στα σχολεία. Και τέλο, ερχόμαι εδώ σε αυτό που είπε ο Ισμαήλ. Προσφυγικά ρεύματα παίζουν και εκεί ένα ρόλο. Αυτά ένα ρόλο. Ποια μπορεί να είναι η επιρροή δηλαδή των προσφυγικών ρευμάτων στην, ε, στα δρομολόγια των σκαφών. Ιδίως εμπορικά σκάφη στην Μεσόγειο διασώζουν πολύ συχνά πρόσφυγες. Δεν έχουν όμως τον κατάλληλο εξοπλισμό. Παίζει κάποιο ρόλο αυτό μέσα στις εργασίες και στις σκέψη σου. Μάριαν Κίλε. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μία ερώτηση να υποβάλω. Έχω να, να υποβάλω μία ερώτηση σε σχέση με την ε, βόρεια διάσταση, δηλαδή της βόρειας αρτηρίας που αφορά τις ε, βόρειες χώρες. Πώς το βλέπετε αυτό ως συντονιστής σε σχέση με τις θαλάσσιες αρτηρίες, γιατί αυτή τη στιγμή ο χάρτης ε, τελειώνει στα νοτιότερα ναι. τμήματα της Φιλανδίας και της ε, Σουηδίας. Τα βορειότερα ούτε φαίνονται. Αλλά εκεί θα βρίσκονται οι μεγάλες αρτηρίες στο μέλλον. Ο Keith Taylor. Δέχομαι και εγώ και πρέπει να τα συγχαρητήρια που εκφράστηκαν και προσχωρώ στο κλαμπ εκείνων που συγχαίρονται τον κύριο Μπράιαν Σίμψον. Ε, Ναι, Δευτέρα, Δευτέρα, Δευτέρα. Monday, Monday, όπως λέει και το τραγούδι. Δύσκολη μέρα. Τι συμβαίνει στον ε, τομέα των θαλασσίων μεταφορών ε, των ε, επιβατών με φέρι και κρουαζιερόπλια και πώς συντονιζόσαστε διασύνοριακά. Τι μπορείτε να κάνετε, τι μπορείτε να προσφέρετε έτσι ώστε και ε, οι επιβάτες να είναι αυτοί που να καρπούνται αυτών των μέτρων. Ε, η κυρία Μοντέιρο Αγγιάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ε, θα δεχτώ αυτά που είπε η κυρία Μάισνερ, ότι όποιος δεν σας ε, γνώριζε θα σας μάθει σίγουρα. Είναι η περίπτωσή μου, γιατί είμαι σχετικά νέα σε αυτό το κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ να μας μιλήσετε για αυτό το λεπτομερές σχέδιο των θαλάσσιων αρτηριών που είναι ύψης της σημασίας για όλους μας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σημεία σε σχέση με τις πράσινες ε, διόδους, τις πράσινες αρτηρίες και την οδηγία σε σχέση με τη χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει η σωστή χρηματοδότηση και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για τη χρήση του LNG, του υγροποιημένου φυσικού αερίου, ως ε, εναλλακτική. Ως προς την ασφάλεια των κρουαζιερόπλειων, θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε καταστάσεις επίγουσας ανάγκης σε σχέση με τα κρουαζιερόπλια και τον τουρισμό στην Ευρώπη. Χαίρομαι γιατί ε, μιλήσατε και για τις πλέον απομακρυσμένες ε, περιφέρειες και τις νησιωτικές περιοχές. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για την Πορτογαλία. Θα θέλαμε να υπάρχει συνδεσιμότητα των νησιών με την Ήπειρο μέσα στα πλαίσια αυτού του ενιαίου ευρωπαϊκού θαλάσσιου χώρου. Θα ήθελα να πω ότι είμαι στη διάθεσή σας για να μιλήσουμε για αυτές τις θαλάσσιες αρτηρίες, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είχα τη χαρά να γνωρίζω τον κύριο Σίμψον γιατί δεν ήμουν στην προηγούμενη θητεία. Όμω διαβάζοντα το έργο ενό ανθρώπου μπορεί να πάρει πολύ ενδιαφέρουσε εικόνε από το περιεχόμενό του. Και η έκθεση πραγματικά κοιτάει σε βάθο τα ζητήματα των θαλάσσιων μεταφορών. Ε, δύο πράγματα μόνο θα ήθελα να πω. Το ένα για την πράσινη ναυτιλία. Ε, τα θέματα τη μείωση των ρήπων της ε, αλλαγής των καυσίμων, της αλλαγής του στόλου σε καινούργια μοντέλα. Είναι όλα πολύ ενδιαφέροντα και όντω και η χρήση του υγροποιημένου αερίου πρέπει να προχωρήσει. Με πολύ ενδιαφέρον είδα πως υπήρχε στην, ε, στο DIP ε, η αναφορά σε ένα σχέδιο που προβλέπει την καθέλκυση συγκεκριμένου τύπου σκαφών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από περισσότερες χώρες σε ευρωπαϊκά ναυπηγεία ε, και με εταιρείε οι οποίε το εξοπλίζουν ευρωπαϊκέ για να μην χρειαζόμαστε να πηγαίνουμε στην Κορέα. Το ερώτημα ήταν, επειδή είχαμε προσπαθήσει να εντάξουμε μια αντίστοιχη ή ε, την, την ίδια προτεραιότητα και στο Juncker Plan, παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν εγγενή προβλήματα στην χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων και αυτό είναι η διαφορά των οικονομιών AAA από τις άλλες οι οποίες έχουν μεγαλύτερο ρίσκο. Και παρατηρούμε ότι όπως και το Juncker Plan μόνο μία ε, επένδυση από την Ελλάδα έχει εγκριθεί, την Ελλάδα που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε. Η χρήση αυτών των εργαλείων το οποίο μας αναφέρατε, πώς θα λάβει υπόψη αυτή την απόσταση που έχουν οι οικονομίες μεταξύ τους ή απλώς θα βοηθάει επενδύσεις που θα γίνονται σε ήδη προχωρημένες οικονομίες. Και το δεύτερο αφορά τις απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές. Ε, στην Αγγλία παραδοσιακά η θάλασσα ήταν αυτό που κρατούσε την ταραγμένη Ευρώπη μακριά. Ε, ελπίζουμε ε, την άλλη εβδομάδα αυτή η απόσταση να μην μεγαλώσει, αλλά για μας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, όπως είναι η Πορτογαλία, η Ιταλία, η θάλασσα ήταν απλώς η προέκταση της ξηράς. Δεν διαφοροποιούσαμε τους δρόμους της θάλασσας από της ξηράς. Βλέπουμε όμως πως στις νησιωτικές μας περιοχές δεν είναι η οικονομική ανάπτυξη η οποία απλώς βελτιώνεται ή μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Είναι η επιβίωση η οποία πρέπει να εξασφαλιστεί. Και πολλές φορές κοιτώντας μόνο το κατά πόσο μία διαδρομή είναι αποδοτική οικονομικά, χάνουμε τελείω τη δυνατότητα να τη στηρίξουμε γιατί αυτή η διαδρομή απλό είναι ο αιμοδότης του νησιού για να μπορέσει να ζήσει και να μην ερημώσει. Πώς λοιπόν και εκεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα μπορέσουν να καλύψουν τέτοιες ανάγκες χωρίς να υποκύψουν σε μια επιλογή η οποία μπορεί να είναι ποιο είναι το πιο ωφέλιμο τελικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Φώστα. Τζάκι Φώστερ, συγγνώμη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και καλώς ήλθες, Μπράιαν, πρώην πρόεδρος. Βεβαίως και μου αρέσει πολύ η έκθεση. Εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών για πολλά χρόνια έχουμε τονίσει τη σημασία του θαλάσσιου τομέα και κάτι που βρίσκω πολύ καλοδαχούμενο είναι την τελευταία δεκαετία ιδίως δηλαδή την εξέλιξη που βλέπουμε και στις εμπορικές μεταφορές και στα επιβατικά πλοία κλπ. Πολύ καλή ιδέα λοιπόν και το γεγονό ότι προωθήθηκε και ε, τελικοποιούνται ας πούμε τα αποτελέσματα. Βέβαια μιας και είμαι από το Λίβερπουλ που είναι βεβαίω ένα από τα κέντρα του κόσμου και με μεγάλη ναυτική ιστορία έχω μια έντονη προσωπική άποψη. Ε, ανακατεύομαι και πάρα πολύ με τα ναυτικά όταν επιστρέφω στην πατρίδα μου. Αυτό που μου αρέσει πολύ είναι το νέο project Ατλαντή. Είμαι βεβαία ότι και η Γαλλία και η Πορτογαλία θα συμμετάσχουν στο έργο αυτό γιατί πρόκειται για λιμάνια στον Ατλαντικό. Και έχουμε και μια ημερομηνία, νομίζω, για την έναρξη, Γενάρη του 17, έναρξη δηλαδή αφετηρία του έργου αυτού. Ρωτώ, Μπράιαν, βρισκόμαστε σε σωστή πορεία και η στήριξη που μπορούμε να δώσουμε, δηλαδή χρηματοδότηση. Έχεις νούμερα σχετικά με τη χρηματοδότηση και πώς μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε. Γιατί μοιραία θα γίνει μεγαλύτερο. Μιλούμε τώρα μονάχα για την αφετηρία ε, στις τρεις πόλεις που προανέφερα. Λιμπεράτσκι. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ πρόεδρε. Φίλε Μπράιαν, όταν σε βλέπω αισθάνομαι ότι επιβεβαιώνεται η άποψή μου ότι υπάρχει και η ζωή και εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί βλέπω να ακτινοβολείς. Χαίρομαι λοιπόν και χαίρομαι που σε βλέπω. Η έκθεσή σου μου άρεσε. Τη διάβασα προσεκτικά και σου δίνω δίκιο σχετικά με το ότι μιλήσε εδώ για short sea shipping και ότι εκεί βλέπεις να διαμορφώνεται ένας ιδιαίτερος βιομηχανικός κλάδος. Το ερώτημα είναι τι υπήρξε πρώτο το αυγό ή η κότα. Αλλά ε, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό. Και αυτά όλα να τα εντάξουμε μέσα στο ευρωπαϊκό μας σύστημα μεταφορών. Και βέβαια πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά και την διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη. Έχω, ας πούμε, να σας κάνω μια σύσταση, να σας δώσω μια συμβουλή. Με αυτές τις θαλάσσιες αρτηρίες μπορούμε να επηρεάσουμε ορισμένες χώρες μέλη, ώστε να βελτιώσουν την πρόσβαση στα λιμάνια. Και από την ενδοχώρα δηλαδή προς το λιμάνι, αλλά και από την θάλασσα και ενώ τις διασυνδέσεις με το σιδηροδρομικό δίκτυο και με, την, με τις γενικότερες μεταφορικές υποδομές στην Ερδοχώρα. Όταν μιλώ εδώ για την Βαλτική, όταν αναλύω την κατάσταση στην Βαλτική, έχω την αίσθηση ότι ακόμα υπολοιπόμεθα πολύ. Στο παράρτημα, ή μάλλον στα παρατήματα 5 και 6, προσπάθησα να βρω τα νούμερα. Για παράδειγμα για πόλεις όπως Ροστόκ, Κουέπελντα, Ντάντσικ. Μάταια όμως έψαξα να βρω το Στετίν και την Γκδίνια. Τα ποσά που βλέπω ανέρχονται σε περίπου 25 εκατομμύρια. Από τα 600 όπως είπες και εσύ. Και μάλιστα και στο παράδειγμα αναφέρεται και ένα ποσό του, της τάξης του 1,4 δις. Άρα είναι πάρα πολύ μικρά τα ποσοστά αυτά. Θεωρείς ότι μπορούμε να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση, διότι εν τέλει έχω την αίσθηση ότι οι κυβερνήσεις και σε αυτές συμπεριλαμβάνω και την Πολωνική δεν έχουν υποβάλει σχέδια για έργα δηλαδή. Θέλουμε μια ενιαία μεταφορική, ένα ενιαίο μεταφορικό χώρο στην Ευρώπη ή όχι. Γιατί εκεί θα παίξει ρόλο και η θάλασσα και οι οδικές μεταφορές. Ευχαριστώ κύριε Νοτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Σίμψον. Δεν είμαι μέλος του φαν κλαμπ σας γιατί δεν σας γνωρίζω. Αλλά ε, θα γνωριστούμε. Κύριε Σίμψον, Είμαι λίγο επιφυλακτική, διότι από το 2001 που συνελήφθη η ιδέα για τις θαλάσσιες αρτηρίες μέχρι σήμερα δεν μου φαίνεται να έχει προχωρήσει πολύ. Και δεν νομίζω να έχουν επιτευθεί οι στόχοι. Το 2001 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πεπισμένη μάλιστα ότι το προϊόν που παρήγαγε τότε θα πρόσφερε μια σημαντική εναλλακτική επιλογή για τις χερσαίες μεταφορές. Πολύ σωστό αυτό οι μεταφορές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός των σύντομων διαδρομών <clears throat> ε, ναυτικών με διαδρομών δηλαδή υπολείπονται κατά πολύ των ε, οδικών μεταφορών, οι, οι θαλάσσιες μεταφορές. Και 2 δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, 400 εκατομμύρια από αυτά προέρχονταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή από την τσέπη του Ευρωπαίου Φορολογούμενου. Αυτά όμω είναι τα χρήματα που έχουν δοθεί και για τη Γαλλία ε, ο απολογισμό δεν είναι και πολύ σπουδαίος. Ε, δηλαδή, Λιόν Τσίτα Βέκια που άρχισε το 2009, καθώ και άλλοι μέχρι το Σαν Ναζέρ που άρχισε το 2010, έκλεισε το 2014, μετά από τέσσερα χρόνια που ε, την εκμεταλλεύτηκαν εφοπλιστές όπως η Γκριμάλντι. Δεν ήταν και πολύ δεν ήταν και πολύ αποδοτική κερδοφόρα η γραμμή αυτή, 21 εκατομμύρια μόνο τον χρόνο, Αποκαταστάθηκε η διασύνδεση αρχές 2015, αλλά για πόσο θα διατηρηθεί ακόμα. Έχετε κάποια ιδέα. Τέλη του 2014 έκλεισε και η διασύνδεση μεταξύ Ζεμπρούκε και Μπιλμπάο, που την χειριζόταν η τρανσφένικα θηγατρική της Ολλανδικής Σπιντόφ. Εάν δεν υπάρξει επαρκής αγορά, οι θαλάσσιες αρτηρίες, δυστυχώς λέω εγώ, θα μείνουν ένα άδειο πουκάμισο, ας το πω έτσι. Δεν θα έχουν μέλλον. και τα χρήματα αυτά και του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου τομέα θα έχουν δαπανηθεί ή μάτιν. Έχουν σημειωθεί και στρεβλώσεις του αγωνισμού από τους μεταφορείς της Ανατολικής Ευρώπης. Έτσι οι θαλάσσιες αρτηρίες δεν μου φαίνονται πολύ αξιόπιστες και πιστέψτε μου, αυτό, πιστέψτε με, αυτό μου φαίνεται ιδιαίτερα λυπηρό. Λοιπόν, ε, ε, αναμένω από εσά να προσπαθήσετε να ανατρέψετε το φαινόμενο αυτό. Ευχαριστώ. Λούση Άντερσον. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω εδώ, Μπράιαν. Συμφωνώ με το Βιμ. Ε, η έκθεση αυτή είναι πολύ μακροσκελής, έχει πάρα πολλά στοιχεία. Ε, μήπως μπορούμε όμως να έχουμε το έντυπο για να το έχουμε και στο γραφείο μας να το μελετήσουμε. Θέλω να κάνω κάποια σχόλια σχετικά με την έκθεση. Το περιβάλλον, όπως είπατε, είναι ύψιστη προτεραιότητα. Προφανώς θέλουμε να αυξήσουμε ε, την, ε, τις καθαρές θαλάσσιες μεταφορές ε, μέσω του project αυτού των θαλασσίων λεωφόρων και να ενισχύσουμε και το οικονομικό ενδιαφέρον για αυτές. Υπάρχει ένα σεμινάριο για τις εκπομπές οξυδίων του αζότου. Αναφέρατε ότι το πλαίσιο το ρυθμιστικό για, τις, ε, για αυτές τις εκπομπές δεν είναι το ίδιο αυστηρό όπως είναι για το άζωτο. Ε, μήπως ε, έχετε κάποια άποψη συγκεκριμένα γι' αυτό, μήπως μπορεί όλο αυτό να ενταχθεί στο μέλλον, στο όλο πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση συνολικά. Και επίσης ένα ακόμα πρόβλημα, βέβαια καταλαβαίνω ότι πλέον η θέση σας δεν είναι πολιτική, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι όλη η συζήτηση για τις εκπομπές και για τις θαλάσσιες μεταφορές και για τη μόλυνση περνάει στην συλλογική συζήτηση που γίνεται για, την, για τον καθαρό αέρα για τις ε, πόλεις, για τα λιμάνια, για τις παραθαλάσσιες περιοχές. Θέλουν να έχουν διάβλους, θέλουν να ανθίσει ή να ανθίσουν θαλάσσιες μεταφορές, αλλά θέλουν καθαρές θαλάσσιες μεταφορές και δεν θέλουν ο αέρας όπως σε, πόλεις όπως ας πούμε ε, το Southampton ή άλλες ε, πόλεις, λιμάνια να μολυνθούν. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και ε, φαντάζομαι ότι θα το κάνετε κι εσείς, οπότε αυτό είναι καλό. Η κυρία Γιάλα Σέντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Μπράιαν στο σπίτι του. Ε, χαίρομαι που σε βλέπω και που χαίρεις άκρα υγείας. Δεν μπόρεσα να διαβάσω το έγγραφο ακόμα, το λάβαμε ηλεκτρονικά, θα το διαβάσω στο εγγύς μέλλον. Είναι γεγονός ότι οι θαλάσσιες αρτηρίες αποτελούν μία πρόκληση και ένα στίχημα για εμάς ως προ τι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Και Σίγουρα θα αυξηθούν οι θαλάσσιες μεταφορές ε, των εμπορευμάτων, διότι είναι πιο εύκολες και λιγότερο δαπανηρές. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω πώς βλέπεις την αύξηση των θαλασσίων μεταφορών εμπορευμάτων αν ε, τελειώσουμε και με τον κανονισμό για τα λιμάνια, πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε το πακέτο αυτό των ε, λιμανιών με τις θαλάσσιες αρτηρίες. Γιατί έχει μεγάλη σημασία να δούμε κατά πόσο θα κινηθούμε προς το καλύτερο ή όχι. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας βοηθήσει η νομοθεσία προς αυτή την κατεύθυνση. Σε σχέση τώρα με τις γειτονικές χώρες, με τη Βόρειο Αφρική και με τη Μεσόγειο, όπως είπε και ο Μπόκουσλαβ για παράδειγμα και ως προς τη Βαλτική, πώς βλέπεις τις εξελίξεις για το ΕΦΣΥ Μιλάμε για την πρώτη αναθεώρηση με τον κύριο Κατάινεν και την ε, ΕΤΕ. Θα μπορούσαμε να έχουμε τομεακές πλατφόρμες για τις θαλάσσιες αρτηρίες, για να είναι πιο δελεαστικές και να έχουμε ένα πιο ολοκληρωμένο δίκτυο με τους λιμένες. Τέλος, ο Κατάινεν μόλις έθεσε τις κατευθυντήριες γραμμές έτσι ώστε το ΕΦΣΙ και τα διαρθρωτικά ταμεία να προβούν σε συνέργειες και θα ήθελα να μας πεις εσύ πώς βλέπεις την συμμετοχή των διαρθρωτικών ταμείων, έτσι ώστε να έχουμε μια καλή χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Τελευταίος ε, μπήκα και εγώ στον κατάλογο των ομιλητών, όπως το έκανες και εσύ πάντοτε, Μπράιαν. Ε, όντως συζητούμε για την μείωση των εκπομπών. Ο, το πιο απλό θα ήταν να έχουμε απαγόρευση και να πάρουμε το ντίζελ. Το ντίζελ βέβαια δεν είναι τόσο καθαρό, αλλά για, με το, σε σχέση με το πετρέλαιο ε, είναι καλύτερο. Είναι τουλάχιστον μια, ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Υπάρχει αυτή η συζήτηση, υπάρχει κάποια τέτοια διάσταση στη συζήτηση. Δεύτερο σημείο. Ξέρω ότι το γνωρίζεις, αλλά με την ε, Επιτροπή μας πήγαμε σε ένα νότιο νησί, ε, το οποίο, και στο οποίο επισκεφτήκαμε έναν λιμένα ο οποίος χτίστηκε με ε, ευρωπαϊκά κονδύλια. Και μάλιστα τα, τόσα χρήματα που κόστησε το λιμάνι αυτό, τα πλοία τελικά δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν γιατί έχει πάρα πολύ αέρα στο λιμάνι. Ουσιαστικά λοιπόν υπάρχει χρηματοδότηση, αλλά οι διάβλοι που υπάρχουν τελικά δεν επωφελούνται. Παρόλο που δαπανώνται πολλά χρήματα. Και άλλο ένα σημείο που θέλω να αναφέρω. Έκανα πρόσφατα μία συζήτηση με μάνατζερ κρουαζιερόπλων και μου ανέφεραν ότι τα κρουαζιερόπλια θέλουν να είναι καθαρά. Υπάρχει αυτό το 0,5% για το 2020, ο στόχος αυτός, και το 0,1% ε, προσπαθούν να το πετύχουν, αλλά θέλουν βεβαίως ε, χρόνο και μας είπαν ότι ε, για τα κροσγερόπλια προσπαθούμε να διαχωρίζουμε τα απόβλητα σε 12 διαφορετικές κατηγορίες. Μιλήσατε πριν για grey water και black water. Grey water είναι αυτό που φεύγει από το ντους ας πούμε και το black water είναι το, το νερό της τουαλέτας. Αυτά όμως μπορούν να, γίνουν, να διαχωριστούν στο λιμάνι. Και ο κανόνας τι λέει, ότι όταν ένα καράβι βρίσκεται 6 χιλιόμετρα μακριά από το λιμάνι μπορεί όλα τα απόβλητα να τα ρίξει στη θάλασσα. Αλλά τα κροσγερόπλια θα πρέπει να ε, επενώνται ή θα πρέπει να αποζημιώνονται με κάποιο τρόπο εφόσον κάνουν αυτό το διαχωρισμό των αποβλήτων. Θα πρέπει κάτι να κερδίζουν από αυτό τον διαχωρισμό. Γιατί δεν φτάνει στην, στον υδροφόρο ορίζοντα των πόλεων. Θα μπορούσε ίσως να χρησιμοποιηθεί αυτό για την παραγωγή ίσως ηλεκτρικού ρεύματος. Αλλά δεν υπάρχει ένα, ή μάλλον υπάρχει μόνο ένα λιμάνι στην Ευρώπη του Αμβούργου που χρησιμοποιείται αυτή η δυνατότητα ηλεκτρικού ρεύματο παραγωγή. Υπάρχει κάτι τέτοιο στο νου σου, κάποιο τέτοιο σκεπτικό. Είναι απλό ουσιαστικά να εφαρμοστεί και για τα κρουαζιερόπλια και για άλλα πλοία για να παραμείνουν όσο πιο καθαρά πράσινα γίνεται. ανεξάρτητα από το πού εκπέμπονται τα αέρια, κάποια στιγμή τα αέρια θα φτάσουν και σε εμά, ακόμα και αν είναι το πλοίο 300 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα. Αυτά από μένα, συνάδελφε Μπράιαν, έχεις το λόγο. He noticed everything, so we let him Okay. Well. Λοιπόν, χαίρομαι που εξακολουθεί να ανθεί ο όμιλος εκτίμησης του Brian Simpson. Για να δούμε τώρα αν θα μπορέσω να απαντήσω και στις ερωτήσεις σας. Δήμ, με ρώτησες για τη βιωσιμότητα και τη δουλειά του IMO. Ναι, συνεργαζόμαστε στενά έχοντας βεβαίως υπόψη ότι ο IMO είναι διεθνής οργανισμός, δεν είναι ευρωπαϊκός, παρακολουθούμε προσεκτικά τι κάνουν, κυρίως για τα θέματα των θαλασσίων, των περιβαλλοντικών συγγνώμη προτύπων. Οπότε ως προς αυτό, προσπαθούμε να πούμε στα κρατημέλη, ας πούμε για τη Μεσόγειο, ότι θα τα καταφέρετε να φτάσετε στο επίπεδο που χρειάζεται. Προσπαθούμε λοιπόν να τα ενισχύσουμε. για, τους, για, τις, την διαφοροποίηση για, τους, ε, για τα είδη μεταφορών. Οι θαλάσσιες λεωφόροι ουσιαστικά είναι η θάλασσα. Αλλά όπως είπα και στους συντονιστές, το θέμα δεν είναι να φτιάξω εγώ ένα ε, υπέροχο κανόνα ο οποίος τελικά να μην μπορεί να εφαρμοστεί πουθενά. Είμαστε λοιπόν σε στενή συνεργασία για να μπορέσουμε να λύσουμε όλα αυτά τα αδιέξοδα, να αποσυμφορήσουμε λίγο τα αδιέξοδα και το πρώτο βήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και το τελευταίο βήμα είναι πολύ σημαντικό για την περαιτέρω πρόθεση των project. Οι εσωτερικές πλωτές ΟΔΗ δεν είναι δικό μου, δική μου αρμοδιότητα, ε, είναι των συναδέλφων μου. Βεβαίως συνεργαζόμαστε στενά για να δούμε τι χρειάζεται. Την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον την προπροηγούμενη εβδομάδα, ήμουν στην Πορτογαλία για, την, ε, για το, και προσπαθούσαμε να δούμε ε, τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Προσπαθήσαμε λοιπόν να, να δούμε κατά πόσο πηγαίνουμε όλοι προς σωστή κατεύθυνση, προς την ίδια μάλλον κατεύθυνση και προσπαθήσαμε να πιέσουμε ώστε να πάμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Τώρα, για την έλλειψη του προσωπικού. Για τα κρουαζιερόπλια συνήθως υπάρχουν κρουαζιερόπλια τα οποία δεν εμπίπτουν στα ευρωπαϊκά, δεν είναι ευρωπαϊκή σημαία. Θα γίνει ένα, μια δοκιμή στη Μάλτα. Νομίζω ότι κάποιος άλλος με ρώτησε γι' αυτό και θα προσπαθήσω να σας πω και άλλα αργότερα για τις υποδομές και τις επενδύσεις σε υποδομές. Πάλι δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, δεν αποφασίζω εγώ ποιες επενδύσεις θα γίνουν, δεν είναι μέσα στην εντολή μου. Αυτό όμως που μπορώ να κάνω είναι να συμφωνήσουμε για project τα οποία μπορούν να ενταχθούν στις προτεραιότητες που έχουμε θέσει. Περιβαλλοντικά, επιμελητία, κατάρτιση κλπ. Αλλά το να κατασκευαστούν ε, ε, γερανοί ε, δεν, είναι, δεν εμπίπτει τουλάχιστον στη δική μου αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες λεωφόρους. Το καταλαβαίνετε φαντάζομαι αυτό. Ισμαήλ. Είναι δύσκολο το θέμα αυτό των θαλασσίων λεωφόρων. Δεν θεωρεί το διάδρομος αρχικά στο τεντή και ούτε καν ε, πολλές φορές ε, σήμερα δεν ε, θεωρείται διάδρομος για το TNT. Αλλά προσπαθούμε να το καταστήσουμε ισότιμο εταίρο. Έχουμε εννέα κάθετους διαδρόμους και δύο οριζόντιους. Ένας από τον οποίο είναι οι θαλάσσιες λεωφόροι. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να προωθούμε το μήνυμα των θαλασσίων λεωφόρων. δηλαδή είναι εξίσου σημαντικές όπως άλλοι. αυτό είναι ο στόχος μας, για να αναγνωρίζει και ο πολίτης ότι οι θαλάσσιες λεωφόροι είναι ένας διάδρομος των TNT. Απλό. Δεν είναι εύκολο βέβαια να γίνει αυτό. Προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Κάτι καταφέραμε, αλλά υπάρχει δουλειά που μπορεί να γίνει ακόμη. Για την διαθεσιμότητα τώρα του LNG, του υγροποιημένου αερίου στα λιμάνια. Μου είπατε για το ε, Αμβούργο. Κάναμε μια μελέτη για το Αμβούργο. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, τα οποία θα τα δείτε και στην έκθεση μάλιστα, που δείχνουν τι είδους ε, κυκλοφορία υπάρχει. Το LNG όμως ε, κερδίζει έδαφος παρά τη χαμηλή τιμή του πετρελαίου. Παρόλα αυτά υπάρχει προτίμηση για το LNG και τη μεθανόλη. Μάλιστα κάποιοι ε, εκπρόσωποι της Σουηδίας από τον Γκέτεμπορκ προσπάθησαν να μετατρέψουν το σύστημά τους να χρησιμοποιεί μεθανόλη και το κάνουν αυτό ε, σε ευρωπαϊκό ε, ταρσανά. Δεν είπαμε ότι θα δοθούν βεβαίω λεφτά εκτό Ένωση. ήταν ευρωπαϊκό ας πούμε το project και τώρα ε, έχουν ξεκινήσει κατασκευή και άλλου σκάφους. Ξεκίνησε λοιπόν έτσι μια κίνια, ένα, μια, ένα ρεύμα και προσπαθούμε να το διατηρήσουμε κινήσει. Βεβαίως παρακολουθούμε το θέμα των προσφύγων. Ακόμα δεν μας έχει δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά οι πρόσφυγες, ε, ουσιαστικά για τους πρόσφυγες μιλάμε για φουσκωτά, οπότε δεν εμπίπτουν ακριβώ στη δική μας αρμοδιότητα, αλλά βεβαίω καταλαβαίνω ότι επειδή είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα φυσικά πρέπει να το παρακολουθούμε στενά. Δεν είναι όμως πρόβλημα αμυγό των θαλασσίων λεωφόρων. Γιατί ξέρετε, κρύβονται σε ρορό, κρύβονται σε κοντέινερ. Ε, είναι λίγο διαφορετικό το πρόβλημα αυτό. Για την ευθυγράμμιση τώρα με το πρόγραμμα. Μάλλον πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω, γιατί στο τέλος τέλος εγώ είμαι η Κομισιόν. Προσπαθώ να, να, να το θέσω διπλωματικά. Καλή ιδέα, αλλά τα λεφτά είναι δικά μας. Τα δικά μας τα λεφτά πήγανε. Οπότε όποιος ε, επανέρχεται Πρέπει να μας πει και τι έγινε τελικά με τα λεφτά αυτά. Για την γεωγραφία τώρα των θαλασσίων λεωφόρων. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί υπάρχουν δύο βασικά project. Η Μεσόγειος και η Βαλτική. Αναμφίβολα η Βαλτική είναι μπροστά από την ε, Μεσόγειο σε ό,τι αφορά τη μεθανόλη, τα εναλλακτικά καύσιμα, το LNG και δεν έχουν και τα απαρχαιωμένα ρορό που υπάρχουν στην ε, Μεσόγειο. Αλλά μελετάτε το θέμα αυτό και από την πλευρά της Μεσογείου και προσπαθεί και η Μεσόγειος να φτάσει τη Βαλτική ως προς αυτό. Η δυσκολία τώρα όμως θα είναι όταν ας πούμε νεολογηθεί ένα πλοίο στην Μεσόγειο πρέπει να πούμε ότι δεν ε, χρειάζεται να επανεφεύρετε τον, τον τροχό. Δεν χρειάζεται να κάνετε από την αρχή μια δουλειά που μπορεί να έχει ήδη γίνει και να έχει αποδεχθεί επιτυχίες. Πρέπει να συντονιστούν λοιπόν τα δύο, να συνεργαστούν οι δύο τομείς σε μια στέρα βάση. Και ελπίζουμε ότι θα γίνει αυτό. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα στις, ε, για τα, στα οποία μπλέκονται, συμμετέχουν τα κράτη της ε, Βαλτικής, στις σκανδιναβικές χώρες. Και μάλιστα ενδιαφέρον ήταν, μάλιστα όταν το έμαθα εγώ, ότι η, η Βαλτική δεν είχε πλήρως μελετηθεί σε γεωγραφική, στη γεωγραφική της έκταση. Έλειπαν κάποια κομμάτια. Υπάρχουν λοιπόν κονδύλια για την διερεύνηση στο, για το σύνολο της Βαλτικής. Η Βαλτική μάλιστα είναι ρηχή θάλασσα και θέλουμε να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Κάναμε μια συζήτηση σήμερα το πρωί η δεν ξέρω όμως κατά πόσο μπορούμε να συντονίσουμε τα πράγματα. Εγώ μίλησα για τις παραμέτρους και για το τι μπορεί να κάνουν κάθε, ο κάθε λιμένας, τι μπορεί να κάνει ο κάθε λιμένας χωριστά. Αλλά αυτό εξαρτάται από το λιμένα για το αν θα υπάρξουν νέα project προγράμματα. Την τελική απόφαση δεν θα την πάρω κατά αναγκή εγώ. Αυτό είναι λίγο ενοχλητικό πρέπει να πω. Τουλάχιστον ενοχλητικό. Δηλαδή μπορούμε να δουλέψουμε ε, εντατικά εμείς, κάποιος να έχει αντίρρηση και τελικά όλη μας η δουλειά να πάει στράφη. Είναι λίγο ενοχλητικό. Δεν το έχω συζητήσει με, τους, ε, με άλλους συντονιστές για να δω αν έχουν το ίδιο πρόβλημα. Δεν το ξέρω αυτό. Για το LNG. Με εξέπληξε εμένα το LNG γιατί θεώρησα ότι οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν στα 48 νομίζω δολάρια του το βαρέλι κάπου εκεί και ότι δεν θα υπήρχε πια η... Δεν θα, μάλλον δεν θα ξεπερνούσαν την ανάγκη να υπάρξει LNG. η Γκριμάλντι λοιπόν που είναι πολύ μεγάλη εταιρεία στη Μεσόγειο ή Στένα στην Βαλτική και άλλη. Ελπίζω αυτές οι μεγάλες εφοπλιστικές εταιρείε να συνεχίσουν λοιπόν να χρησιμοποιούν το υγροποιημένο φυσικό αέριο στα πλοία τους. Τα Μάικλ, Τα βρώμικα νερά. Ναι, καλύτερα να διάζονται, να γίνεται η εξεργασία τους δηλαδή, η κατεργασία τους, στο λιμάνι. Αλλά πρέπει να ασφαλίσουμε ότι το λιμάνι θα διαθέτει την απαραίτητη υποδομή για να δέχεται τα χρησιμοποιημένα τα βρώμικα νερά. Κοιτάζουμε λοιπόν να φτιάξουμε προγράμματα στήριξης για να μπορούν τα πλοία να αποχετεύουν εκεί τα βρώμικα νερά τους. Τώρα, εκπαίδευση. Ναι, είμαι και συντονιστής για την εκπαίδευση. Ανησύχησα πολύ διότι πήγα σε ορισμένα λιμάνια και είδα ότι προσπαθούν να φτιάξουν ένα κλάδο κουραζιέρας. Εδώ μιλάμε για κουραζιερόπλια που υποδέχονται 5.000 άτομα και με τρία τέτοια κουραζιερόπλια, τρία ή τέσσερα μέσα στο λιμάνι σου, στην περίπτωση της Μάλτας για παράδειγμα, είναι περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι κατοικούν στη Βαλέτα. Ρώτησα λοιπόν τι είδου σχέδια έχουν αν κάτι πάει άσχημα. Η Μάλτα, ειλικρινώς, οι άνθρωποι μου είπανε δεν έχουμε σχέδια. Και αποφάσισαν λοιπόν να κάνουν μια άσκηση στη διάρκεια της δικής τους προεδρίας όπου να γίνει ας πούμε μια εκένωση ενός κρουαζιερόπλου κάτι τέτοιο. Τα ίδια στην Ισπανία με χρήση των υπηρεσιών κατεπίγουσας ανάγκης γαλλικών και ισπανικών κάναμε το, την άσκηση αυτή και πήγε πολύ καλά. Έχουμε λοιπόν γνώση του τι γίνεται εάν κάτι πάει άσχημα στην περίπτωση ενός κουραζιρόπιου, αν και Ευχόμαστε ποτέ να μην γίνει τίποτα το άσχημο, έτσι. Αλλά πρέπει βέβαια να σχεδιάσει κανείς και για την αντιμετώπιση μιας επίγουσας κατάστασης. Δεν είναι βέβαια μονάχα περιπτώσεις όπως η Κώστα Κονκόρδια. Μπορεί να ξεσπάσει μια επιδημία, μια νόσος του λεγιοναρίου ε, λόγω του νερού κτλ. μέσα στο σκάφος. Υπάρχουν αρκετές κλίνες στα νοσοκομεία για να φροντίσουν τους ανθρώπους κτλ. Τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι για τη μετανάστευση απάντησα ήδη. Τώρα, η Nordic Dimension, η βόρεια διάσταση. Συμφωνώ μαζί σας ότι η διαδρομή από τη Βόρεια Θάλασσα δεν έχει μπει τόσο πολύ ακόμα επιτάπητος. Θα μπει όμως. Οι θαλάσσιες αρτηρίες ε, δεν φτάνουν μόνο μέχρι το Λίβερπουλ, και πάνε και μέχρι τον Ατλαντικό. Κάνουμε λοιπόν το σχετικό σχεδιασμό και η Northern Sea Route θα ενταχθεί και αυτή. Για την ώρα είναι στη φάση του σχεδίου, γιατί βεβαίως παίζει ένα ρόλο και η Ρωσία. Και ε, μιλεί για, μάλλον για τον Northern Sea Passage ο Brian Simpson, που είναι άλλο πράγμα. Ε, πάντως, χαίρομαι που μίλησες γι' αυτό, για την Nordic Dimension, γιατί χρειάζεται και υπηρεσίες παγωθραστικών που είναι πολύ σημαντική στην περίπτωση αυτή και κανένας δεν το κατανοεί στην Ευρώπη. Ο Κύπριος υπουργό να κοίταξε με τεράστια απορία όταν του μίλησε για τα φιλανδικά παγωθραστικά που όμως είναι σημαντικό όπλο για να μένει ανοιχτή η θαλάσσια οδός στη Βαλτική το χειμώνα και βέβαια ελπίζω και το βόρειο πέρασμα. Περνάει δηλαδή από την Αρκτική. Γιατί είναι αυτή η Σουηδία, όχι ναι, Φιλανδοί. Ε, φιλανδικά παγωθραστικά λοιπόν έτσι. Θα χρειαστεί να παίξουν ένα ρόλο και αυτά. Keith, Keith Taylor. Αυτό το short sea shipping έχουμε ξοδέψει πολλά λεφτά για την ανάπτυξη και το short shipping και τα οχηματαγωγά roll-on, roll-off τα εξετάζουμε για την ενδεχόμενη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Όταν μιλούμε τώρα όμως για ασφάλεια, εκπαίδευση κλπ. δεν μιλάμε μονάχα για κουραζιερόπλια, μονάχα για το Βασίλισσα Βικτωρία ή το Βασίλισσα Ελισάβετ αλλά και τα οχήματα ογά, ρολών, ρολόφ και και όλα τα ζητήματα ασφάλειας που άπτονται αυτών. Δεν είναι τόσο έντονα τα πράγματα εκεί, διότι ε, τα πληρώματα είναι από Ευρωπαίους πολίτες. Ωστόσο χρειάζονται εκπαίδευση και αυτή και χρειάζεται να εκπαιδευτεί το πλήρωμα και για τη χρήση των διάφορων μέσων κλπ. ώστε να γνωρίζουν πολύ καλά τι πρέπει, τι έχουν από κάτω τους τέλος πάντων όταν κινούνται διασχίζοντας ε, το κανάλι της μάχης ή οτιδήποτε άλλο. Μα ούτε τα μισά δεν έχω πει ακόμα, πρόεδρε, για την Πορτογαλία. LNG πάλι νομίζω ότι είναι το καύσιμο του μέλλοντος. Δεν λέω ότι και καλά πρέπει οπωσδήποτε να είναι το LNG. Άμα είναι καθαρό, ναι. Άμα είναι καθαρό καύσιμο, βέβαια. Αλλά σήμερα κυρίως το LNG είναι αυτό που προσφέρει καθαρό. Για τα τα είπα, η σύνδεση περιφερειακών περιοχών, τα είπα αυτά στην ομιλία μου, εσένα σκεφτόμουν άλλωστε, είναι σημαντικά αυτά για μένα. Όπως έχουν τα πράγματα τώρα, οι θαλάσσιες αρτηρίες συνδέουν βασικά λιμάνια μεταξύ τους. Εγώ θέλω να αλλάξει λίγο αυτό. Κεντρικό λιμάνι, κόπορ, δηλαδή με άλλα λιμάνια, σύνδεση με άλλα λιμάνια, γιατί και υπάρχουν και άλλα σημαντικά λιμάνια που έχουν και διασύνδεση με την ενδοχώρα πλέον. Κύριος, κύριος Κύρκος, ο κύριος Κύρκος, συγγνώμη. Νέα τεχνολογία, νέα σκάφη, νέα ναυπηγεία, είπα κάτι σχετικά. η προσέγγιση γεωγραφικών περιοχών. Όπως έλεγα στον Κλοντ, πρέπει να δεις με την θαλάσσια μεταφορά στην εξωτερική περιφέρεια και πώς αυτά θα προσεκίσουν το κέντρο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και βέβαια μέσα στα πλαίσια των κανόνων που έχουμε για την ώρα. Τζάκι, εσύ. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε έχει αναγνωρίσει τη σημασία του ναυτιλιακού τομέα. Δεν ξέρω αν άλλοι έχουν αντιληφθεί. Και το Liverpool Atlantic Project. Ναι, βεβαίως και είναι μέσα στο σχεδιασμό μας. Μπόγκουσλαφ. Α, έφυγε. Short Sea Shipping. Και συνοχή. Κοιτάξτε, παιδιά, προσέξτε. όταν δόθηκε η συνοχή στις χώρες μέλη, όλες εκτός από μία την Ελλάδα χρησιμοποίησαν τη συνοχή για τις θαλάσσιες αρτηρίες. Όλες οι άλλες χρησιμοποίησαν για τους σιδηρόδρομους. Εγώ δεν είμαι αντίθετο με τους σιδηρόδρομους, έτσι ο Μάικλ Κράμερ, αλλά δεν ενδιαφερόταν καθόλου να χρηματοδοτήσουν τις θαλάσσιες αρτηρίες. Και μόνο με τη δική σα βοήθεια μπορέσαμε, δηλαδή μπορέσατε να πείσετε τις κυβερνήσεις των χωρών μελών σας, ώστε κάποια, κάποιες από τις χρηματοδοτήσεις για τη συνοχή να πάνε και στις θαλάσσιες αρτηρίες. Το Στετίν δεν το βρήκε. Να του πει κάποιος ότι η πολωνική κυβέρνηση δεν υπέβαλε σχετική αίτηση. Μαρή Κριστίν. Δεν θα σου πω ότι δεν επιδοτούμε τους δρόμους και τις διαδρομές μάλλον και το 2010 ήταν πρόγραμμα Μάρκο Πόλο και όχι το πρόγραμμα των θαλάσσιων αρτηριών. Αν είσαι παράπονα, στο Μάρκο Πόλο. Δεν επιδοτούμε τις διαδρομές λόγω της πολιτικής ανταγωνισμού. Δεν μπορούμε να δώσουμε σε μία διαδρομή λεφτά σε βάρος μιας άλλης. Δεν τα κάνουμε αυτά. Συμφωνώ ότι οι θαλάσσιες αρτηρίες έχουν ξεκινήσει με δυσκολία. Αλλά δεν συμφωνώ μαζί σου ότι δεν οδηγούν πουθενά. Προχωρούν κάπου και τελικώς, όπως λένε στα αγγλικά, τη δοκιμάζεις την πίτα στο τέλος όταν θα ε, τη Εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι τελικά θα υλοποιηθούν. Και το βλέπεις και στο γεγονός ότι έχουμε τέσσερις φορές παραπάνω αιτήσει για έργα που έχουμε λάβει. Λούσι Βαριά καύσιμα. Άλλη υπόθεση αυτή. Νομίζω ότι πρέπει να περιληφθούν. Μίλησα και στην αρχική μου μιλία. Α, ξέχασα τώρα ακριβώ τι είπα. Αλλά είπα τέλο πάντων καθαρό ατμοσφαιρικό αέρα. Και αυτό είναι, αυτός είναι ο στόχο μα. Οι νιές αύξηση των θαλάσσιων μεταφορών. Όπως είπα και πριν, θα δούμε στο τέλος. Αλλά επαναλαμβάνω ότι 40% του εσωτερικού εμπορίου, 40%, 4-0, 40, γίνεται με τα καράβια, με θαλάσσιες μεταφορές. Αλλά βέβαια δεν το ακούμε αυτό, διότι, κοιτάξτε, τα εμπορευματοκιβώτια δεν ψηφίζουν οι νέες. Μακάρι, μακάρι να ψήφιζαν. Και γι' αυτό δεν ακούμε πολλά σχετικά. Είπε όμως κάτι σωστό. Τρίτες χώρες. Έχουμε κάποια έργα σε συνεργασία με τρίτες χώρες. Έχουμε τα νοπά προϊόντα με Παλαιστίνη και Ισραήλ. Επίσης η διασύνδεση με το Μαρόκο. Και βγαίνοντας στον Ατλαντικό ελπίζω να αποκατασταθούν περισσότερες διασυνδέσεις και με τη Βόρεια και Νότια Αμερική, χρησιμοποιώντας το Ατλαντικό τόξο. Και για τις εσωτερικές υδάτινες διαδρομές, αντιλαμβάνομαι την απογοήτευση της Κάρλας για τον Δούναβη. Και Μιχαήλ εσύ, Κράμπερ το βαρύ δίζελ, το δίζελ γενικά. Εγώ θέλω να φύγω από το βαρύ καύσιμο για προφανείς λόγους. Αποφυγή τώρα ε, <laughs> λιμανιών που έχουν ισχυρούς ανέμους. Καινούριο στοιχείο αυτό. Τι να το κάνεις σε ένα λιμάνι άμα δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Ε, ε, λιμάνι για παράδειγμα στο βορρά που είναι αποκτισμένο 11 μήνε το χρόνο από του πάγου. Πρέπει να το δούμε βέβαια όταν θα σκεφτούμε πού θα χρηματοδοτήσουμε. Για Blackwater είπαμε ε, ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε ένα έργο το, το οποίο στηρίζουμε διαμήκους της Βαλτικής ένα ηλεκτρικό οχηματαγωγό. Κάνουμε την προσπάθειά μας και εμείς. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το αναπτύξουμε, να το εξελίξουμε. Για ε, διαχείριση κρουαζιερόπλειων τα είπα. Ε, θα πρέπει βέβαια να συμπαραταχθεί μαζί μας ολόκληρος ο κλάδος των κρουαζιερών. Αν ξέχασα κανέναν, ελπίζω όχι. Πάντως νομίζω ότι απάντησε όλους. Αγαπητέ Μπράιν, νομίζω ότι απάντησες σε πολλές ερωτήσεις δέχθηκες και πολλές, πολλές φιλοφρονήσεις. Όταν ήσουν πρόεδρος δεν θυμάμαι να σου κάναν τόσες πολλές φιλοφρονήσεις. Πάντως, πολύ χαρήκαμε που σε είδαμε, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε για όλα. Και θα σε ξαναδούμε το αργότερο την επόμενη εβδομάδα. Θα σας δω ορισμένους βεβαίως στο Ρότερνταμ την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή σας, καλή τύχη και θα ξανάρθω σε 12 μήνες για να σας πω πώς πάμε. Ελπίζω και εσείς να συμβάλλετε με τις δικές σας εισρωές μέχρι τότε. Ευχαριστώ και πάλι. So, wir bleiben im Grunde bei dem Thema zur Freisetzung des Potenzials der Λοιπόν, ε, πάμε στην απελευθέρωση του δυναμικού για τις ε, ιστορικές ε, οδούς, ε, για, την, για τις παράκτιες περιοχές και συμβολή στην πολυτροπική μεταφορά επιβατών. Ο Keith Taylor είναι ο εισηγητής. Έχεις το λόγο, Keith. Well, hi. Thank you much. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ένα λεπτό να ησυχάσουν όλοι. To continue because of the time. Σας παρακαλώ πρέπει να συνεχίσουμε. Αν θέλετε μπορείτε να αποχωρήσετε. Okay, well, thank you, Chair. I think that uh, everybody is leaving silently. Um... Όλοι βλέπω ότι αποχωρούν. Χαίρομαι για τη δυνατότητα που μου δίνεται σήμερα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί μέχρι τώρα για τις παράκτιες περιοχές και τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις μεταφορές ολοκληρωμένα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες. Χαίρομαι γιατί μπορέσαμε να συνεργαστούμε πολύ καλά με τους σκιώδεις. Ε, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ότι τα οχηματαγωγά πλοία μπορούν να μας βοηθήσουν για μια ε, βιώσιμη πολιτική μεταφορών. Γι' αυτό ε, ασχολήθηκα με την ασφάλεια, διασυνοριακή συνεργασία, περιβαλλοντικές προδιαγραφές και αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, καθώς και τα δικαιώματα των επιβατών. Πολλοί, όπως ξέρουμε, ε, μεταφέρονται οδικά, δηλαδή ακολουθούν σε οδικές αρτηρίες και αυτό δημιουργεί μεγάλες στενοπούς. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να προωθήσουμε τη μεταφορά μέσω πλοίων για να έχουμε και καλύτερες υπηρεσίες μεταφοράς. Επίσης, ε, να αποφύγουμε τις ε, στενοπούς και τη συμφόρηση και τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα. Γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις εσωτερικές πλωτές οδούς, την ακτοπλοεία και τη θάλασσα. Και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερες μεταφορές, πιο οικονομικές και περισσότερη ευημερία για την προστασία και του περιβάλλοντος της Ευρώπης. Η μεταφορά των επιβατών έχει μεγάλη σημασία και στην ακτοπλοεία και γι' αυτό χρειαζόμαστε στατιστικά στοιχεία για τις πλωτές μεταφορές. Ιδιαίτερα σε σχέση με τις θαλάσσιες υπηρεσίες ως προς τις φορτηγίδες, τα κρουαζιερόπλια και ούτω καθεξής. Μας ενδιαφέρει επίσης να λάβουμε υπόψη την ικανότητα μεταφοράς, ε, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού. Και μέσα στα πλαίσια των δημοσίων μεταφορών, πιστεύω ότι τα απορθμία μπορούν να προωθήσουν την ποιότητα ζωής προστατεύοντας το περιβάλλον. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο οι πλωτές μεταφορές μπορούν να βελτιστοποιήσουν το τουριστικό δυναμικό ε, φέροντας σε επαφή και απομακρυσμένες περιοχές μέσα στα πλαίσια των ε, πολυτροπικών μεταφορών. λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα όλων των επιβατών, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν περιορισμένη κινητικότητα, καθώς και τους τουρίστες. Μιλάμε για 400 δις που ε, διαπλέουν τα τα, τις θάλασσες και φτάνουν στα λιμάνια μας. Και γι' αυτό θα πρέπει αυτά τα 15 χρόνια να δούμε πώς, μπορούμε, πώς ανταποκριθήκαμε και πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε και για αποφυγή ατυχημάτων. Και φυσικά και για να προωθήσουμε τη διάσωση των ανθρώπων. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη συμμόρφωση με τα κοινά ευρωπαϊκά ε, πρότυπα ασφαλείας, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τους υπάρχοντες κανόνες και να προωθήσουμε και τις ε, καινοτόμες ε, τεχνολογίες να προωθήσουμε την αιωλική ενέργεια, την ηλιακή, τα εναλλακτικά καύσιμα και ούτω καθεξής στον τομέα μεταφορών, καθώς ε, και αποδοτική χρήση της ενέργειας. Γι' αυτό το ε, Interreg, το EFSI, το CEF και άλλα μέσα είναι τα καταλληλότερα προς την ε, κατεύθυνση αυτή. Συνάδελφοι, εύχομαι να συνεργαστούμε στο εγγύς μέλλον για την έκθεση αυτή. Ο Σαλατόρ Πολιέζε έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, διάβασα με μεγάλη προσοχή αυτό το σχέδιο γνώμης, σχέδιο έκθεσης και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τέιλορ γιατί προσπαθούμε να ενισχύσουμε αυτό τον τομέα μεταφορών που για γεωγραφικούς και μορφολογικούς λόγους είναι ύψης της σημασίας. Σημερίζομαι την ανάγκη διατροπικών μεταφορών και ενίσχυσής τους. Και φυσικά και την μεταφορά των επιβατών και εναερίως, παράλληλα με τις μεταφορές εμπλό, μέσα στα πλαίσια των δημοσίων δικτύων και φυσικά και να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος. Επίσης, συμμερίζομαι την ανάγκη βελτίωσης της ασφάλειας μέσω της κατάρτισης του προσωπικού. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί ένας τέτοιος νέος οργανισμός ή να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας, τους φορείς που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Ο κύριος Κύρκος έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Τέιλορ, για το ολοκληρωμένο σχέδιο που μας παρουσίασε. Μπορώ να συμφωνήσω με τη γενική προσέγγιση του ότι πρέπει να ενισχυθεί η χρήση των οχηματαγωγών για τους λόγους που πολύ σωστά μας περιέγραψε σήμερα. Θα ήθελα να επισημάνω μόνο τα παρακάτω σημεία. Καταρχάς πρέπει να γίνει ξεκάθαρος ο διαχωρισμός μεταξύ οχηματαγωγών και κρουαζιεροπλοίων. Ο τίτλος της έκθεσης αναφέρεται μόνο στα πρώτα, αλλά στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα κρουαζιερόπλαια που έχουν όμως άλλη δυναμική, άλλες δυνατότητες, άλλες απαιτήσει, άλλο κέντρο βάρους, κυρίως επειδή τα κρουαζιερόπλαια αποτελούν μέσω αναψυχής, ενώ το χηματαγωγά μέρος της καθημερινής μεταφοράς φορτίων και επιβατών. Δεύτερο, θεωρώ ότι ιδιαίτερο βάρο πρέπει να δοθεί στην υποβοήθηση των περιφερειακών και παραμεθόριων περιοχών, όπω είπαμε και στην προηγούμενη κουβέντα μα, ελληνικά νησιά, Μαδέρα, Αζόρε, Κανάρια, δεν μιλάμε για ανάγκε τουρισμού ή μεταφοράς κάποιων προϊόντων, μιλάμε για επιβίωση όλων αυτών των περιοχών που χωρίς το χηματαγωγά δεν μπορούν. Οπότε πρέπει να εξασφαλίσουμε με όποιον τρόπο γίνεται δωδεκάμινη ε, δράση των δρομολογίων. Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εντοπίσει διαφορετικά τι προκλήσει σε διαφορετικέ περιοχέ. Άλλε είναι ανάγκε τη Βαλτική, όπου εκεί πρέπει ίσω να μιλήσουμε για περισσότερα και καινούργια δρομολόγια πορθμίων, και άλλε τη Μεσογείου, όπου βρίσκεται περισσότερο από το ίμιση του στόλου και των υπηρεσιών, και εκεί θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε στην αναβάθμιση των οχηματαγωγών πλοίων. Σημαντική επίση αναφορά πρέπει να γίνει για τη σύνδεση με την ενδοχώρα των λιμένων που εξυπηρετούν τα οχηματαγωγά πρέπει να αναφερθούμε και στον τομέα των σιδηροδρόμων και των οδικών μεταφορών και στην πρόσβαση εσωτερικής ναυσιπλοείας στους λιμένες, αν θέλουμε να αυξήσουμε την πολυτροπικότητα. Στι αστικές περιοχές τα πορθμία πρέπει να είναι μέρος της πολυτροπικότητας, που σημαίνει πιο ολοκληρωμένα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων και τους χρόνους επιβίβασης κλπ. Τελειώντα, θα ήθελα να πω ότι με βάση και τα τελευταία δεδομένα πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα για την ασφάλεια των επιβατών, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην εμποδίζουν με κανένα τρόπο την ομαλή ροή τόσο των επιβατών όσο και των εμπορευμάτων. Έχει αποδειχθεί ότι η συνεργασία των, των υπηρεσιών και η πρόληψη είναι πολύ πιο αποδοτική από του σκληρού και χρονοβόρου ελέγχου. Τέλο, αξίζει να σημειωθεί ότι από τότε που αρχίσαμε να εργαζόμαστε σε αυτό το σχέδιο, η Επιτροπή έχει υποβάλει νομοθετικέ προτάσει για την επικαιροποίηση των υφιστάμενων οδηγιών, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων για την ασφαλή λειτουργία των οχηματαγωγών πλοίων, καθώ και νομοθεσίε για την ασφάλεια των επιβατικών πλοίων. Είμαστε σίγουροι πω αυτή η έκθεση πρωτοβουλία θα βοηθήσει και την επερχόμενη δουλειά μα σε αυτού του φακέλου. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Vielen Dank. Jetzt ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Κίθ για την έκθεσή σου. Καλό είναι που ασχολούμαστε τώρα με το θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι όντως ε, πολύ καλό που θέλεις ε, να προωθήσεις τα ρορό και τα οχηματαγωγά και τα φέρει, που ούτως άλλως είναι ένας πολύ καλός, ε, ένα πολύ καλό μέσο μεταφοράς. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε βιώσιμες ε, μεταφορές, βεβαίως πρέπει να προωθήσουμε τις ιστορικές πρώτες μιλάμε για επιβάτες, είτε μιλάμε για ε, εμπορεύματα, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την ε, συμφόρηση ή να αποσυμφορήσουμε λίγο τις χερσές μεταφορές. Επίσης είναι πολύ σημαντικό, όπως είπαν και πολλοί συνάδελφοι, η σύνδεση των νησιών με την ενδοχώρα και ταιριάζει όλο αυτό και στα πλαίσια των θαλασσίων λεωφόρων Βεβαίω δεν μπορούμε να χρηματοδοτούμε παντού και τα πάντα που θα το ήθελαν οι πολίτε, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Ένα σημείο που θέλω να υπογραμμίσω και έχω την ίδια άποψη με τον ε, εισηγητή για τα ε, Είναι πραγματικά τεράστιο ε, ε τομέα ανάπτυξη. Εκεί μπορεί να ενταχθεί και η πτυχή τη ε, κινητικότητα. Ε, οι αδερφοί μου με τον γαμπρό μου πήγανε μια ε, κρουαζιέρα και ίσω σε ε, να μπορεί κανείς να κάνει κρουαζιέρα και σε ποτάμια ε, κάποια στιγμή. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε αν θέλουμε περισσότερα πλοία, αν θέλουμε να έχουμε όντω πλοία θέλουμε περισσότερο ε, έμπειρο προσωπικό και καταρτισμένο, πρέπει να, τα πλοία μας να είναι καθαρά, πρέπει να δούμε τι κάνουμε με τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και τέλος θέλουμε να έχουμε καθαρές θάλασσες, καθαρούς ποταμούς. Προφανώς αυτό εντάσσεται και στην μπλε ανάπτυξη. Πρέπει να επικεντρωθούμε λοιπόν και σε αυτό. Και ε, να πω επίσης ε, ε εξοπλισμό των ε, λιμένων. Βεβαίως μιλήσαμε και για τον Blackwater πιο πριν, για τα λίματα, για την επεξεργασία τους. Και αυτό θα πρέπει να, γίνεται, να μπορεί να γίνεται σε όλα τα λιμάνια. Πρέπει λοιπόν και εκεί να στοχεύσουμε την προσοχή μας. Και επίσης προτάθηκε να υπάρξει μια ειδική υπηρεσία. Ναι, τα... Εμένα με ενδιαφέρουν πολύ τα θαλάσσια θέματα. Καλό ακούγεται να έχουμε αυτή την υπηρεσία, αλλά πάντα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όταν φτιάχνουμε νέε δομέ διοικητικέ, γιατί πρέπει ε, να δούμε τα τις αρμοδιότητες που θα έπαιρνε αυτή η νέα υπηρεσία αν μπορούμε να τις δώσουμε στις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες και να μην φτιάξουμε άλλο ένα επίπεδο γραφειοκρατίας. Αυτά από μένα και ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεση. Ευχαριστώ. Η κυρία Νοτιού. Merci, Monsieur le Ευχαριστώ. Το σχέδιο είναι γενικά καλό. Έχουμε ορισμένες επιφυλάξεις. Ξεκινάμε από την ε, διαπίστωση ότι θα πρέπει να εντατικοποιηθεί αυτή η μορφή μεταφοράς και είναι η πλέον καθαρή. Η Κομισιόν δεν είχε προωθήσει μία ολοκληρωμένη μελέτη χρηματοδότησης από τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ένας ενιαίος χώρος μεταφοράς δια των πλωτών οδών και ίσως χρειάζεται και ένας ευρωπαϊκός οργανισμός εσωτερικής ε, ναύση πλοίας. Ίσως βεβαίως βάζουμε ένα νέο φόρτο με έλεγχους και ίσως θα πρέπει να υπάρξει και μία τυποποίηση προς τα κάτω, ιδιαίτερα για την προστασία των επιβατών. Ας μην γίνει ένα επιπλέον θέμα το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος ε, ενδελεχώς και εις βάθος, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι τα μη ορυκτά καύσιμα είναι πανάκια για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν πρόκειται για μία μαγική ράβδο. Θα πρέπει τα δικαιώματα των κρατών μελών να ισχύουν και σε αυτή την εσωτερική ναυσή πλοία και η μεταφορά με φέρει θα πρέπει να ε, διευκολυνθεί. Ε, ξέρω κύριε Τέιλορ ότι είσαστε Βρετανός από τον Χάρι Πότερ, αλλά δεν έχετε μαγικό ραβδί. Ο κύριος Καραμίτσος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ τον εισηγητή και όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν εδώ Είναι η πρώτη προσπάθεια που γίνεται και στην τελική έκθεση θα ε, υποβοηθήσουμε και εμείς για να σας δώσουμε πληροφορίες και στοιχεία, επιπρόσθετα στοιχεία. Λοιπόν, μερικά σημεία που θα ήθελα να θίξω. Καταρχήν, Μιλάμε για την κοινή πολυτροπική χρήση ε, οχηματαγωγών ε, πλοίων για τη μεταφορά και επιβατών. Δηλαδή έχουμε τις ε, μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών. Μιλάμε για ένα 95% που είναι συνδυασμένες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών. Δηλαδή δεν έχουμε μία αμυγή μεταφορά επιβατών. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και για τις μελλοντικές δράσεις. Ως προς την ασφάλεια των επιβατών θα πρέπει να γνωρίζετε ότι την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίναμε τρία μέτρα που κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση Καταρχήν η καταγραφή επιβατών. Θυμόσαστε ε, πέρσι το μεγάλο ατύχημα μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας όπου χρειάστηκαν τρεις εβδομάδες για να δούμε ε, πόσοι ήταν οι αγνοούμενοι. Γι' αυτό προτείνουμε βελτίωση σε αυτό το τομέα της καταγραφής επιβατών. Επίσης την προώθηση ε, προδιαγραφών ασφαλείας για τα οχηματαγωγά πλοία στην εσωτερική πλοία μέσα στα πλαίσια του Ρίφιτ και επίσης τα οχηματαγωγά στις ε, τακτικές γραμμές. Πιστεύω ότι αυτά τα τρία στοιχεία θα ε, μας ε, κρατήσουν αρκετά δραστήριους φέτος και του χρόνου μέσα στα πλαίσια και του έτους θαλασσίων μεταφορών. Ως προς την περιβαλλοντική πλευρά υπάρχουν ε, ε, πολλά θέματα που μας απασχολούν μέσα στα πλαίσια των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και θέλουμε η ευρωπαϊκή νομοθεσία να αντικατασταθεί από μία διεθνή απόφαση που συζητείται αυτή τη στιγμή στον IMO και να φτάσουμε σε μία συμφωνία και με τους ευρωπαϊκούς φορείς και μετά θα γίνει και η κατάλληλη προσαρμογή. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να τονίσω πέρα από το περιβαλλοντικό είναι η γενικότερη πολιτική μας. Αν θυμόσαστε υπάρχει αυτή η θαλάσσια στρατηγική και έχουμε πέντε συνιστώσεις δηλαδή την ασφάλεια, τη θαλάσσια ασφάλεια και την ψηφιοποίηση και απλούστευση του πλαισίου μεταφόρων. Επίσης, τη βελτίωση του short sea shipping, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και εναρμόνιση και ίσως μπορούμε να έχουμε περισσότερο input. Ένα άλλο θέμα είναι οι μεταφορές μας, οι θαλάσσιες μεταφορές να γίνουν πιο ανταγωνιστικές διεθνώς, με βάση τις αποφάσεις σε διεθνές επίπεδο και ένα πέμπτο σημείο, το οποίο θέλουμε να τονιστεί ιδιαίτερα, είναι τα επαγγελματικά προσόντα των εργαζόμενων στις θαλάσσιες μεταφορές, διότι ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους νέους, οι οποίοι πολλές φορές έρχονται για να εργαστούν στον τομέα του short sea shipping, αλλά μετά αποθαρρύνονται γιατί το 40% των μεταφορών ανήκει στο, στους Ευρωπαίους. Είναι πλειοκτήτες και μεταφορείς. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το προσωπικό αυτό χρησιμοποιεί την πείρα του και την ε, διαθέτει, τη διαδίδει. Είμαστε στη διάθεση του εισηγητή για να συνεργαστούμε περισσότερο γιατί η Επίτροπος θα σας πει αργότερα πώς έχει σημασία μέσα στα πλαίσια του έτους θαλασσίων μεταφορών να συνεισφέρουμε και να εμπλουτίσουμε αυτό τον τομέα. Γιατί έχει σημασία να δούμε και τα, το εναχόμενο κόστος των θαλασσίων μεταφορών, αλλά ως προς το short sea και το διεθνές κομμάτι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση. Ιδιαίτερα για αυτούς που εργάζονται στον ένα τομέα και μεταβαίνουν στον άλλον. Εδώ θα παραμείνω γιατί θα μπορούσα να συνεχίσω, μιλάω για το ΣΕΦ, το ΤΕΝΤΗ, καθώς και τα δικαιώματα των επιβατών και την χρηματοδότηση των σχεδίων. Αλλά δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας, θα μπορέσουμε όμως να συνεργαστούμε με τον εισηγητή για να δούμε ποια στοιχεία θέλει να συμπεριλάβει στην έκθεσή του. Και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο λειτουργίας. Ευχαριστώ. Κιθ, ως εισηγητής λαμβάνεις πάλι το λόγο. Η τελευταία λέξη, έτσι είναι. Λοιπόν, Ευχαριστώ όλες και όλους για την καλή υποδοχή που επιφυλάξατε στην έκθεση και εσείς οι σκιώδεις ιδίω. Σημειώνω τα σχόλιά σας. Σημειώνω επίσης ότι αρκετοί από εσά εκφράσατε για κάποια ανησυχία για την νέα πρόταση για ένα νέο οργανισμό εσωτερικών υδάτινων οδών. Αυτό πρέπει να αναπτυχθεί και να συζητηθεί. Υπάρχει, είναι ελκυστικό το να υπάρξει μια συνεκτική προσέγγιση από τον οργανισμό. Δηλαδή, μάλλον τα καθήκοντα του οργανισμού αναλαμβάνουν τώρα διάφοροι άλλοι φορεί μέχρι τώρα. Κάτι τέτοιο λοιπόν μπορεί να συζητηθεί και περισσότερο. Η αναγνώριση επίσης των πρόσθετων πλεονεκτημάτων που μπορούν να σφέρουν οι υδάτινες μεταφορές και ιδίως η δυναμικότητα, ή μάλλον η δυνατότητα που προσφέρουν να μειωθεί η, η υπερβολική πυκνότητα των αστικών κέντρων. Και βέβαια είναι και πολύ ευχάριστο να ταξιδεύει κανει ε, από τη θάλασσα. Ε, αναφέρθηκε η Επιτροπή και στην εκπαίδευση. Σήμερα το πρωί άλλωστε μιλήσαμε για τα επαγγελματικά προσόντα των ε, όσων ασχολούνται με την εσωτερική ναυσιπλοεία με τους εμπειρογνώμονες και με τους συναδέλφους. Τα συζητήσαμε αυτά. Ε, ο συνολικός στόχος της έκθεσης είναι να διευκολύνει ευφιέστερα και, και, και πιο πράσινα ταξίδια, πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Ε, και αυτές τέτοιες προτάσεις θα κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 23η έκτου στις 12 το μεσημέρι. Τελειώνει εδώ η συνεδρίαση της Επιτροπής. Συνεχίζουμε τώρα με τους συντονιστές ή αν θέλετε και κλεισμένο των θυρών ώστε θα περιμένω να εγκαταλείψουν την αίθουσα όσοι δεν έχουν το δικαίωμα να παρίστανται.